χαιρετήσω και μια αντιπροσωπεία από την Ελβετική Ομοσπονδία που βρίσκεται στα θεωρία και χαιρετίζω τον πρόεδρο του Ελβετικού Εθνικού Συμβουλίου. και τους άλλους βουλευτές οι οποίοι είναι παρόντες από το Ελβετικό Εθνικό Συμβούλιο. Υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι σε, ως μέλη διαφορών επιτροπών είχαν την ευκαιρία ήδη να συζητήσουν με τους συναδέλφους μας από την Ελβετία και να συζητήσουν για θέματα των μελλοντικών σχέσεων Ελβετίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός ο διάλογος φυσικά θα συνεχιστεί και στο μέλλον και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας αγαπητοί συνάδελφοι από την Ελβετική Στομοσπονδία. Ψηφοφορίες τώρα. Ξεκινούμε με την έκθεση Γκρόμπαρτσικ σε σχέση με τα αποθέματα Σολομού στην